Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε. Δεν κατάλαβα καν πώς πέρασε η ώρα. Πήγε ήδη και 25. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους ε, που είναι παρόντες. θα ξεκινήσουμε, μεταδίδεται και στο διαδικτύο συνεδρίαση περίεργο σήμερα το πρωινό λόγω και της απεργίας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε πάντες. Θα ακούσουμε την παρουσίαση της κυρίας Βασιλιάδου που είναι ο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και καλωσορίζω σε αυτή την κοινή συνεδρία των δύο επιτροπών και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ισότητας των Φίλων. Και καλωσορίζω θερμότατα την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΦΑΜ, την κυρία Χάνιμπολ, ε, είμαστε και στην ίδια εκλογική περιφέρεια και όλος τυχαίω σήμερα είναι και η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που είμαστε ευρωβουλευτέ που συμπροεδρεύουμε σε τη επιτροπής. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την εξάλληψη του τράφικινγκ της εμπορίας ανθρώπων που αποκαλείται η στρατηγική ήταν το, ο κύριος μηχανισμός για την ανάπτυξη, συντονισμό και εφαρμογή των ευρωπαϊκών δράσεων στον τομέα αυτό. Σε προηγούμενα ψηφίσματα και των δύο επιτροπών επισημαίνουμε το, τον ιδιαίτερο τροτό χαρακτήρα που έχουν και το πόσο ευάλωτοι είναι στο τράφικινγκ οι αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, και μετανάστε και τονίσαμε την ιδιαίτερη προσοχή που θα πρέπει να δοθεί σε γυναίκε παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδε και ζητούμε αυξημένη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών στα ψηφίσματά μα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι συνέχεια έχει δοθεί στη στρατηγική και κυρίως πόσε στοχευμένε προτεραιότητε συμβάλλουν στην αναβάθμιση των ευρωπαϊκών προσπαθειών να αποτραπεί, να προληφθεί η εμπορία ανθρώπων. Θα δώσω το λόγο πρώτα στη Μέρι Χάνιμπολ, που είναι αντιπρόεδρο τη Επιτροπής ΦΑΜ, για να κάνει κάποια σύντομα εισαγωγικά σχόλια και να παρουσιάσει ε, την κυρία Βασιλιάδο που θα μας κάνει την ενημέρωση ω συντονίστρια κατά του τράφικινγκ. Όπως ε, είπε, Κλώδη, είναι η πρώτη φορά που έχουμε την τύχη να συμπροεδρεύουμε, ενώ και, ήδη, ε, και οι δύο εκλεγόμαστε στο Λονδίνο. Και ακριβώς είναι σημαντικός ο λόγο που ασχολούμαστε με το τράφικινγκ γιατί σίγουρα είναι το Λονδίνο προορισμός ε, τέτοιας εμπορίας ανθρώπων. Και το θέμα αυτό μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές και μας απασχολεί ιδιαίτερα και στην Επιτροπή ε, των γυναικών ε, προβληματιζόμαστε για το θέμα αυτό, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες και κυρίως για σεξουαλική εκμετάλλευση. Εδώ, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΦΑΜ, είμαι συμπρόεδρος αυτής της κοινή συνεδρίασης και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά του συμμετέχοντε. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι το θέμα της εμπορίας ανθρώπων είναι πολύ σημαντικό και όλο και περισσότερα θύματα υπάρχουν. Ε, πολύ περισσότερα από αυτά που δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Και η συντριπτική πλειοψηφία, όπως είπαμε, είναι γυναίκες και κορίτσια που γινόνται θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ε, σωματεμπορίας. Και δεν νομίζω ότι αυτό το στοιχείο ε, συγκεντρώνει τη δέουσα προσοχή μέχρι στιγμής. Γι' αυτό και θα πρέπει από εδώ και πέρα να λαμβάνετε πολύ περισσότερη υπόψη στις ευρωπαϊκές στρατηγικές, ε, τα σχέδια δράσης που υιοθετούμε και τα μέτρα που υιοθετούμε για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Και τώρα με ιδιαίτερη χαρά να δώσω το λόγο στην κυρία Βασιλιάδου που είναι η συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και έχει συμβάλει τα μάλα ε, στην προσπάθεια καταπολέμησης αυτής της μάστιγας και θα μας παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την εξάλληψη του τράφικινγκ της εμπορίας ανθρώπων και θα μας παρουσιάσει και τις ε, περαιτέρω συγκεκριμένες δράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ε, δύο προέδρους των Επιτροπών Λίμπε και ΦΑΜ για την πρόσκληση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν ε, θερμός υπέρμαχος ε, και ε, προσιλωμένος σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον αγώνα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Για να διευκρινίσω, έχουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την εξάλληψη του, της εμπορίας ανθρώπων για την περίοδο 2012-2016 και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε όλους τους στόχους και να υλοποιήσουμε όλους τους στόχους της προηγούμενης στρατηγικής και τώρα μετά από αξιολόγηση του νέου γεωπολιτικού πλαισίου ε, θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις και τις προτεραιότητες μας για την επόμενη περίοδο. Δεν είναι μια στρατηγική καθ' αυτή, αλλά ένα σύνολο φιλόδοξων δράσεων ε, και αξιών που θα διέπουν το έργο μας. Ήδη παρουσιάσαμε την ανακοίνωση αυτή στα κράτη-μέλη και στην κοινωνία των πολιτών και έχουμε λάβει μέχρι στιγμής πολλά θετικά σχόλια για τις προτάσεις μας και ευχαριστώ τους ενδιαφερόμενους για τα σχόλιά τους. Ε, το όλο έγγραφο της ανακοίνωσης περιστρέφεται γύρω από την πρόληψη, γιατί οτιδήποτε άλλο εμφανίζεται κατόπιν εορτή για τα θύματα οποιασδήποτε μορφή εκμετάλλευση. Οπότε εμά αυτό κυρίω μα ενδιαφέρει, η πρόληψη. Και αυτό αναφέρεται ρητά και στην οδηγία του 2011 για την ε, καταπολέμηση του τράφικινγκ, ότι η θεμελιώδη σημασία έχει η πρόληψη. Επίσης, ενώ η εμπορία ανθρώπων είναι μια πολύ επικερδή δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματο, ταυτόχρονα συνιστά και μια κατάφορη παραβίαση ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνεται και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί οριζόντια, γιατί συνδέεται με πολλές ε, πολιτικές. Επίσης, αυτό αναγνωρίζεται και στην ανάλυση της Europol για την αξιολόγηση απειλής για σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Τη συνιστά σημαντική δηλαδή απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εμπορία ανθρώπων. Αυτό αναφέρεται επίσης σε πολύ σημαντικά έγγραφα που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως το θεματολόγιο για τη μετανάστευση, για την ασφάλεια. Αυτά είναι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και στο θέμα της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Περνώ κατευθείαν στους ε, λόγους ε, που διέπουν το έργο μας. Ήδη αναφερθήκατε στη διασύνδεση με τη μετανάστευση. Βέβαια, η εμπορία ανθρώπων δεν είναι ε, φαινόμενο της μετανάστευσης. Δύο τρίτα, μάλιστα, των θυμάτων είναι Ευρωπαίοι υπήκοοι. Αυτό μας λέει ε, η ευρωπολα από τα περσινά στοιχεία και από την ε, Eurostat επίσης τα στοιχεία συνηγορούν προς αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα όμως να πω κάτι που έχουμε Το 2016 η Διεθνή Οργάνωση για τη Μετανάστευση εντόπισε 11.000 γυναίκες και κορίτσια που έφτασαν από τη Λιβύη ή από την Ιγυρία μέσω της Λιβύης στη Ρώμη. Και 80% αυτών είναι θύματα ε, σωματεμπορίας, δηλαδή 9.000 από τις 11.000 μόνο στο 2016, μόνο ε, σε μία χώρα, μόνο μέσω Λιβύης προς τη Ρώμη και μόνο μέσα σε ένα χρόνο. Τόσα πολλά θύματα και αν υπολογίσουμε τα κέρδη των ε, εμπόρων μόνο για το 2016 9.000 θύματα, σκεφτείτε, 10 με 20 πελάτες τη μέρα, 5 με, 9, 99 ε, ευρώ ανά σεξουαλική εκμετάλλευση και ε, σχεδόν όλες τις μέρες του χρόνου. Έχουμε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δισεκατομμύριο κέρδη μόνο από σεξουαλική εκμετάλλευση, χωρίς καν να λαμβάνετε υπόψη ε, το νόμιμο κέρδος των νόμιμων επιχειρήσεων και των ε, νόμιμων επιχειρήσεων που αποκομίζουν παράνομα κέρδη. Έχουμε 9.000 ε, γυναίκες και κορίτσια που κάπου ε, στεγάζονται, κάπου τρώνε, κάπου μετακινούνται και χρησιμοποιούν διάφορες υπηρεσίες. Μερικοί το γνωρίζουν, άλλοι όχι. Μερικοί φορές είναι συνειδητοί η εκμετάλλευση, άλλες όχι. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλε τι πτυχέ αυτή τη αλυσίδα εμπορία ανθρώπων. Και αυτό και είναι ο τίτλο τη πρώτη προτεραιότητα. Για ένα 12χρονο κορίτσι σε ένα χωριό στην Ιγυρία να καταλήξει στι Βρυξέλλε. Σκεφτείτε πόσοι, έχουν, πόσοι μεσάζοντες, πόσοι καταχραστές, πόσοι εγκληματίες ή και πόσοι που ακούσει συμμετέχουν στη διαδικασία ή ερήμην του χωρί να γνωρίζουν την κατάσταση και με πόσου μεσάζοντε έχουν επαφή αυτά τα θύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ε, εξαρθρώσει αυτή την αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων και να κόψει αυτούς τους κρίκους αλυσίδας. Για όλες τις ε, νεαρές γυναίκες και για τα κορίτσια που είναι μέσα στα 9.000 θύματα του 2016, σκεφτείτε τους δράστες της ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ας πούμε 5 με 20 ε, πελάτες τη μέρα, μόνο για ένα χρόνο, μόνο για 350 μέρες το χρόνο, μόνο για 9.000 κορίτσια. Δεν θέλω καν να κάνω τους μαθηματικούς υπολογισμούς. Και ούτε ένας δράστης δεν έχει διωχθεί, δεν έχει ε, καταδικαστεί από ό,τι ξέρουμε ή στο, στο μέτρο που θα θέλαμε. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τους, τις προσπάθειές μας παρεμπόδιση του επιχειρηματικού μοντέλου αυτών των ε, εγκληματικών δικτύων και κυκλωμάτων. Και επίση θέλουμε να θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη, τα μισά τουλάχιστον κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το έχουν κάνει, να ποινικοποιήσουν αυτού που συνειδητά χρησιμοποιούν υπηρεσίε θυμάτων εμπορία ανθρώπων. Και πραγματικά αυτό που με σοκάρει είναι ότι πολλέ χώρε-μέλη όταν κάποιος έχει συνείδηση της κατάχρησης και ότι χρησιμοποιεί με τον ΑΒ τρόπο ε, κάποιο θύμα του εγκλήματος αυτού και παρόλα αυτά δεν τον ενοχοποιούν ή δεν ποινικοποιούν αυτή τη συνειδητή χρήση αυτής της υπηρεσίας. Γιατί μπορεί κανείς ε, να αγοράσει παράνομα ένα προϊόν και να ε, διωχθεί, αλλά όταν αγοράζει ε, παράνομα την ε, υπηρεσία ενός θύματος τράφικινγκ μπορεί να μην είναι Θέλουμε λοιπόν να ε, δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ευθύνης Έχουμε το άρθρο 23.2 της οδηγίας του 2011 και θα πρέπει να δοθεί μια συνέχεια για να ποινικοποιούνται τέτοιες συμπεριφορές. Η οδηγία ζητά από τα κράτη-μέλη να ποινικοποιήσουν τέτοιες συμπεριφορές, δηλαδή εκείνους που συνειδητά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός θύματος ε, εμπορίας ανθρώπων. Η οδηγία βέβαια προσπαθεί να θεσπίσει κάποια ελάχιστα πρότυπα και προδιαγραφές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη όχι μόνο σκεφτεί, αλλά δεν έχουν ποινικοποιήσει τέτοιες συμπεριφορές. Αυτό που συνειδητά δηλαδή ε, εμπλέκονται σε ένα τέτοιο έγκλημα. Επίσης, όπως είπα, θα πρέπει να μεριμνήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε κάθε μηχανισμό για να βοηθήσουμε και να θαρρύνουμε τις ε, ε, δημόσιες αρχές να να διαταράξουν αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο με μεθοδολογίες, με επιχειρησιακές δραστηριότητες, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να διεξαγάγουν έρευνες, να διώξουν τους δράστες, να δημιουργήσουμε ικανότητες, να αναπτύξουμε μηχανισμούς και εργαλεία και κυρίω κάτι που το έχω ζητήσει επανειλημμένα στα κράτη-μέλη, να συστήσουμε κοινέ ομάδε ερευνών, όχι μόνο εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τρίτε χώρε. Η εμπορία ανθρώπων έχει πολλές μορφές. Η κυρία Χάνιμπολ πολύ σωστά είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια και κυρίως για σεξουαλική εκμετάλλευση. Πέραν τούτου όμως έχουμε και άλλα θύματα για εργασιακή εκμετάλλευση. Και αυτό θα πρέπει να σταματήσει όχι μόνο εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παντού στον κόσμο. Είναι λοιπόν προτεραιότητά μα να προθεωρήσουμε βιώσιμε επιχειρηματικέ πρακτικέ και αξιοπρεπεί εργασιακέ συνθήκε στι χώρε παραγωγή με πολλού και διάφορου τρόπου, αλλά κυρίως να εξασφαλίσουμε ε, αλυσίδες εφοδιασμού και αξιών που δεν θα περιέχουν και ε, εμπορία ανθρώπων. Και αυτό τα λέμε στην ανακοίνωση. Δυστυχώ γνωρίζουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερα θύματα και γνωρίζουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει εργαστεί εκτενώς ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν τα νομοθετήματα εκείνα που θα προστατεύουν τα θύματα. Το πρόβλημα είναι ότι η νομοθεσία και η εφαρμογή αυτής. Το να εξασφαλίσει κανείς ότι τα θύματα πράγματι ασκούν τα δικαιώματά τους. Επιδιδόμαστε λοιπόν σε μια σειρά από δραστηριότητες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας και τους οργανισμούς μας για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουμε αυτή την άσκηση των δικαιωμάτων. Και ε, πρώτη προτεραιότητα, όπως έχει ζητήσει η Επιτροπή Γυναικών, βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ισότητας των Φύλων για να δοθεί υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη, προκειμένου αυτά με τη σειρά τους να υποστηρίξουν τα ε, θύματα. Και επίσης ε, κατευθυντήρες γραμμές που έχουμε εκδώσει για την αποτροπή ε, τη, του, της εμπορίας ε, παιδιών και ανθρώπων ευρύτερα βρισκόμαστε σε μια ε, διαδικασία βεβαίως προστασίας των, ε, των ανθρώπων. Ε, ξεχνούμε όμως κάποιες φορές ότι ε, τα δύο τρίτα των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων είναι Ευρωπαίοι πολίτες και παιδιά. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση αυτό. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να προσδιορίζουν, να εντοπίζουν τα θύματα. Βλέπουμε τους μηχανισμούς εντοπισμού των θυμάτων, εκπονούμε σχετικές μελέτες και θα εκδώσουμε και καθετήριες γραμμές συμβουλές προς τις εθνικές αρχές για τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων. Και εδώ θέλω να πιστήσω την προσοχή σας γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε επανειλημμένως. Έχουμε ε, ένα, μια σειρά από προβλήματα όπως είναι η, η σύγχρονη δουλεία, η καταναγκαστική εργασία, η παιδική εργασία, Βάζουμε όλα αυτά μέσα στον ίδιο κουβά. Είναι πολύ βολικό βεβαίως ε, ε, αν κανείς είναι δημοσιογράφος ή πολιτικός, αλλά καθόλου βολικό ε, δεν είναι αυτό για τα θύματα που δεν προστατεύονται από τον νόμο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ορισμούς από την νομοθεσία, έχουμε το πρωτόκολλο του Παλέρμου, αυτά είναι τα εργαλεία για την προστασία των θυμάτων. Πρέπει να λογοδοτήσουμε, είμαστε υπόλογοι και απέναντι στα θύματα και πολλά κράτη-μέλη λοιπόν έχουν ζητήσει να υπάρξει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια γύρω από αυτές τις ε, έννοιες. Και κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και συγκεκριμένα της, ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θέλουμε να ε, ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επιδόμαστε και σε αυτό το έργο κατόπιν ετήματος και του Ελληνικού συνεδρίου και με βάση και τους στόχους για το 2030. Ε, πολλές φορές ε, ε, ιδίως όσον αφορά τον επικεντρωνόμαστε στον βιώσιμο στόχο για την καταπολέμηση της, της καταναγκαστικής εργασίας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι 80% των θυμάτων, γυναίκες και παιδιά, εμπίπτουν σε έναν στόχο που τείνουμε να αγνοούμε. Και εδώ κάνω έκκληση στην Επιτροπή σας να κάνουμε ε, ίσες προσπάθειες για την επίτευξη και των τριών στόχων για την καταπολέμηση του τράφικινγκ σε όλες τις μορφές του. Επίσης, ε, βρισκόμαστε σε συνεργασία με, τις, με, τις, με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ε, στον τομέα της δικαιοσύνης και, της, ε, και των εξωτερικών υποθέσεων. Ήταν, έχει εκδοθεί και μια σχετική ανακοίνωση, ήταν εξαιρετικό το έργο αυτό. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι περισσότεροι οργανισμοί θα δραστηριοποιούνται και θα συνεργάζονται στον τομέα αυτό και συνεργαζόμαστε βεβαίως με την, την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ που μεταξύ άλλων έχει ως στόχο την καταπολέμηση του τράφικινγκ. Ε, θέλω να σας... Έρθω στα υπόλοιπα της εξωτερικής διάστασης, αλλά θέλω να διαβεβαιώσω ειδικά την Επιτροπή Γυναικών πως αυτά τα ζητήματα αφορούν άμεσα την εξωτερική διάσταση του ζητήματος της ισότητας. Ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα για το τράφικινγκ, να καταλάβουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Οπότε δημοσιεύσαμε μία μελέτη όχι μόνο για το οικονομικό κόστος, το οποίο είναι τεράστιο αστρονομικό και δεν ξέρουμε πού πάνε τα κέρδη, αλλά και για το κοινωνικό και ανθρώπινο κόστος. Και πάλι, σεβόμενοι τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου σε ένα ψήφισμα, θα δημοσιεύσουμε μία μελέτη για τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την ε, καταπολέμηση τη διακίνηση για σεξουαλική εκμετάλλευση και για την διάδοση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών τη Ένωση. Ε, ναι, τελειώνω. Και θα δημοσιεύσουμε την επόμενη έκθεση προόδου σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγία, όπου τα κράτη-μέλη θα στείλουν στη συντονίστρια εμένα δηλαδή εμπροκειμένο τα αποτελέσματά τους και εμείς θα συντάξουμε μια ευρωπαϊκή έκθεση και θα ε, δημοσιεύσουμε τα δεδομένα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλα τα κράτη-μέλη που έχουν στείλει τα δεδομένα τους. Τέλος, θα ξεκινήσουμε μια πανευρωπαϊκή καμπάνια ενημέρωσης ε, για την ε, παράνομη διακίνηση ανθρώπων και αυτό θα γίνει μέσω της στήριξης των στόχων καταπολέμησης της σωματεμπορίας σε διάφορα προγράμματα και υποτεραιότητες όπου υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Το κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και ακριβώς για να ανταποκριθούμε στις ε, δεσμεύσεις μας και τις υποχρεώσεις μας ε, θα δούμε το τι πρέπει να γίνει από πλευράς ασύλου, ασφάλειας, ε, πρόσβαση δικαιοσύνη, προενταξιακή κινητικότητα και τα λοιπά. Για να τελειώσω το σημαντικότερο θέμα ε, που το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε την εφαρμογή και τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του κοινοτικού δικαίου. Ξανά και ξανά έχω πει ότι έχουμε εξαιρετική νομοθεσία και αυτό οφείλεται βεβαίω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα έχει πενιχρά αποτελέσματα αν δεν εφαρμοστεί σωστά. Οπότε η δουλειά της ε, Κομισιόν είναι να κάνει αυτό ακριβώς ε, και αυτό κάνουμε και δεν θα διστάσουμε να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την συντονίστριά μας. Συνάδελφοι, έχουμε ψηφοφορία στις 12, κάτι το οποίο είναι γελίο, γιατί πρέπει να γίνει η συζήτηση σε 15 λεπτά. Αντάσου ε, αν θα προσπαθήσουμε. Αν μπορείτε να περιοριστείτε σε δύο λεπτά, παρακαλώ, συνάδελφοι. Ξέρω βεβαίω ότι σας απογοητεύει, αλλά προσπαθείτε να... προσπαθήσετε. Λοιπόν, Κριστίν Ρεύο πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βασιλιάδου. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας που πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Η οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορία ανθρώπων φυσικά θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Το είπατε και εσείς στα συμπεράσματά σας. Στη συζήτηση στο Στρασβούργο τον περασμένο Ιανουάριο, ο, κύριο, ο Επίτροπος Αβραμόπουλος μας είπε ότι οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζουν το βαθμό μεταφοράς στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας. Θα πρέπει να είναι αυστηρή και προσεκτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εν ανάγκη να, ξε... γύρει και διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, διαδικασίες επιπαραβάση κατά των κρατών μελών. Επίσης, να ζητηθεί συνεργασία και με άλλες χώρες. Όπως είπατε, είναι δισεκατομμύρια τα κέρδη των εγκληματικών κυκλωμάτων της εμπορίας ανθρώπων. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ των χωρών μελών για τα οικονομικά θέματα. Επίσης, ε, καλές οι δηλώσεις, αλλά καλύτερη στρατηγική. Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα φαινόμενο που συνεχίζεται και μάλιστα οξύνεται και σίγουρα τα επίσημα στοιχεία υποτιμούν την πραγματική κατάσταση. Θα πρέπει να έχουμε μια συγκρίσιμη μελέτη μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που προποθέτει εναρμόνιση των δικτών και των ορισμών. Έχω τρει συγκεκριμένε παρατηρήσει. Καταρχήν, τα θύματα τη εμπορία ανθρώπων θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια παραμονή, ακόμη και αν δεν μπορούν να συνεργαστούν με την αστυνομία. Ε, με ανησυχούν κυρίως ε, οι μετανάστριες, γυναίκες και κορίτσια. Επίσης, ο σχετισμός της εμπορίας ανθρώπων με άλλες παραβάσεις, όπως το λαθροδιακίνηση μεταναστών. Επίσης, θα πρέπει να θεσπίσουμε μια ανθρωπιστική βίζα, ώστε να μπορούν να φτάνουν ε, με ασφάλεια στα σύνορα, χωρίς να επιχειρούν επικίνδυνες μεταβάσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά που είναι και τα πιο ευάλωτα. Επίσης, πριν από 15 μέρες πήγα στη Γαλλία σε ένα κέντρο υποδοχής Όλες οι γυναίκες στο κέντρο αυτό είχαν υποστεί τουλάχιστον μια φορά βιασμό κατά τον περίπλο τους ε, προς την Ευρώπη. Επίσης, ε, ε, θα πρέπει να καταργηθεί το μέτρο της διοικητικής κράτης, όπως ισχύει δυστυχώς. Επίσης, να παράσχουμε ψυχολογική βοήθεια σε αυτά τα θύματα και φυσικά ποινική βοήθεια Ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά την συντονίστρια για το πολύ αποτελεσματικό της έργο. Ευχαριστώ κυρία Βόζεμπερκ. Πρόεδρε, καταρχάς να συγχαρώ τη Μύρια τη Βασιλιάδου για το πολύ σημαντική δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Το γεγονός ότι επισκέπτεται κράτη-μέλη αλλά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνει και προσπαθεί να συντονίσει προσπάθειες αυτό το οποίο μας απασχολεί, ε, συνάδελφοι, σήμερα και το οποίο εντάσσεται και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στην Επιτροπή ΦΑΜ, όπου έχω την τιμή να μετέχω, μας έχει ευαισθητοποιήσει σε πάρα πολλές συζητήσεις. Όμως βρισκόμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί μέχρι στιγμής να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Και αυτό διότι αυξάνεται το φαινόμενο και εμείς έχουμε βήματα πίσω. Τι θέλω να πω με αυτό. Η οδηγία η οποία, την οποία καλούμαστε να εφαρμόσουμε ως εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών, σε πρώτη κατεύθυνση πρέπει να έχει εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, έτσι ώστε ενιαία να αντιμετωπίζεται. Βέβαια αυτό εντάσσεται στην κατασταλτική ε, οπτική του φαινομένου. Στην προληπτική που πολύ σωστά έβαλε έμφαση και η κυρία Βασιλιάδου έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι οργανωμένα τα κράτη-μέλη στις υπηρεσίες τους, στην ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σε συντονισμένες προσπάθειες που να εμπλουτίζουν τις υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, διότι όλοι ξέρουμε, είναι κάτι που δεν δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση, ξέρουμε ότι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και που τροφοδοτεί αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις κυρίως και πρωτίστως γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Εκεί λοιπόν κάθε κράτος μέλος που έχει πολύ συγχρονισμένες και συντονισμένες προσπάθειες της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος μπορεί να συμβάλλει σημαντικά. Συμφωνώ τέλος με την κυρία Βασιλιάδου για μια ευρωπαϊκή καμπάνια η οποία θα ενημερώνει για την έκταση του φαινομένου στα κράτη-μέλη αλλά νομίζω ότι επίσης πρέπει πρέπει να δώσουμε έμφαση στη συνεργασία των κρατών μελών με τις τρίτες χώρες όπου έχουμε στα πλαίσια της μετανάστευσης και του προσφυγικού πολλά θύματα του τράφικινγκ και κάνω διάκριση ιδιαίτερα στην σεξουαλική ε, εκμετάλλευση των θυμάτων αυτών η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες αλλά είναι και αγόρια. Ξέρουμε ότι το φαινόμενο έχει πλέον ε, ε, δεν έχει έμφυλα χαρακτηριστικά, αφορά και στα δύο φύλλα και σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός και ο συντονισμός των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των ειδικών υπηρεσιών και η δική μας συνεργασία σε νομική εξέλιξη του νομοθετικού φαινομένου νομίζω ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank ευχαριστώ συνάδελφοι. Ο κ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ πως ε, πραγματικά αξίζει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή. Εσείς πώς ε, το βλέπετε, πώς θα μπορούσε να διαδοθεί η γνώση για το θέμα αυτό σε ένα ευρύτερο κοινό. Τι θα πρέπει πραγματικά να γίνει πολύ πιο γνωστό πέρα από αυτή την αίθουσα για να αντιληφθεί ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και έχω και άλλη μία ερώτηση. Πώς εκτιμάτε το κλείσιμο της ε, Βαλκανικής ε, οδού σε σχέση με το θέμα μας έχει οδηγήσει σε μείωση της εμπορίας ανθρώπων ή τι ακριβώς συνέβη. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Χιμένεθ, παρακαλώ για δύο λεπτά. Θα προσπαθήσω ούτε δύο λεπτά, γιατί βιάζομαι κιόλας. Αυτό που θα ήθελα πρώτα απ' όλα είναι να συγχαρώ εκ βάθους καρδίας την κυρία Βασιλιάδο για το θάρρος της, ε, την τόλμη της, την αφοσίωσή της, ε, την πραγματική της προσήλωση στο θέμα, τον ενθουσιασμό και το ζήλο που έχει δείξει, που έδειξε και συνεχίζει να δείχνει. Και θα ήθελα να τη συνδράμω και να πω ότι συμμεριζόμαστε τον εκνευρισμό της ε, και την ανησυχία της, γιατί πραγματικά δεν φαίνονται πάντα τα αποτελέσματα, γιατί μερικές φορές πρέπει να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία και την παθητικότητα των κρατών μελών, που δεν χορηγούν τα στοιχεία που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δεν εφαρμόζουν τις συστάσεις. Και αυτό που είπατε στο τέλος είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχουμε καλή νομοθεσία για τα θύματα, αλλά αν δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτή, αν δεν ενημερώνονται τα θύματα, αν υπάρχει άγνοια και στα θύματα και στους δικαστές και στην αστυνομία, αν δεν γίνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης, τότε δεν βοηθάμε, παρά την καλή νομοθεσία που έχουμε. Και στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει έχουμε το ίδιο παράδειγμα ε, με την ψηφοφορία που θα έχουμε στις 12. Καλή νομοθεσία, αλλά καλύτερη εφαρμογή. Επίσης, ε, τα θύματα είναι ίδια. Δεν υπάρχουν καλύτερα θύματα και χειρότερα θύματα. Όλοι έχουν τα ίδια αισθήματα. Αλλά δεν έχουν όλα τα θύματα τις ίδιες ανάγκες. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να βάζουμε όλα τα, τα θύματα στο ίδιο τσουβάλι. Άλλο ένα θύμα τρομοκρατίας και άλλο ένα θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή εργασιακής εκμετάλλευσης. Κάθε θύμα ανάλογα με τις ανάγκες του θα πρέπει να τύχει διαφορετικής προστασίας και θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση γιατί τα κράτη-μέλη βάζουν όλα τα θύματα στο ίδιο τσουβάλι κάτι που αποβαίνει βάρος τελικά του συμφέροντος των θυμάτων. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Βασιλιά ε, για την ε, δουλειά σα και για τα αποτελέσματα που έχετε στο στο αυτό ζήτημα. Έχω δύο ερωτήσει, Ναι, συμφωνούμε όλοι ότι είναι θέμα όχι μόνο νομοθεσίας ε, από πλευράς κοινοβουλίου στο θέμα του ποινικού δικαίου που κάναμε ένα μεγάλο βήμα, αλλά βεβαίως θα πρέπει ακριβώς να υπάρχει ένας αντίκτυπος στην πραγματικότητα. Για να γίνει αυτό όμως έχει σημασία να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η διάσταση του φαινομένου, ειδικά για την σεξουαλική εκμετάλλευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς έχει κατάσταση στο κάθε κράτος μέλος. Έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Ακριβή δεδομένα. Μια χαρτογράφηση δηλαδή της σχετικής ε, μαφίας. Ε, γιατί έχουμε τη διέστηση ότι το φαινόμενο είναι τεράστιο στην Ισπανία και στην Ιταλία, αλλά ξέρουμε ακριβώς την ε, διάσταση σύμφωνα στην κάθε χώρα. Και η άλλη ερώτηση είναι, έχουμε μια χαρτογράφηση επίσης των βέλτιστων πρακτικών. Δηλαδή, να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφοριοδότες σε τέτοιες ε, ποινικέ ε, περιπτώσεις ε, περιπτώσεις διακίνησης ανθρώπων να λαμβάνουν υπηκότητα, να λαμβάνουν προστασία νομική για όσους αποκαλύπτουν τέτοια κυκλώματα. Αυτό νομίζω θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ε, ξέρουμε λοιπόν ποιε είναι οι καλές ε, πρακτικές ε, που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη για την ώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κιέγγε, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Κλοντ. Και εγώ είχα να υπογραμμίσω κάποια πράγματα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πραγματικά πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Πρώτα απ' όλα, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι οι πρέπει να έχουμε δεδομένα ασφαλή, έγκυρα που αφορούν όλες τις μορφές ε, βίας. Είτε είναι σεξουαλική ε, βία, αλλά υπάρχει και μια άλλη πτυχή η οποία αφορά το λαθρεμπόριο οργάνων. Πάρα πολλά παιδιά, νέοι έχουν, ένα, έχουν χάσει ένα όργανο και θεωρώ ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται. Ειδικά στους ανήλικους περνάει σχεδόν απαρατήρητο. Το άλλο θέμα είναι οι πόροι. Οι πόροι που πρέπει να διατηθούν στα κέντρα κατά της ε, βίας που στηρίζουν τα θύματα και συντονίζουν τον αγώνα κατά της ε, βίας εις βάρος των γυναικών. Και η διαδικασία ένταξης. Η ένταξη είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ε, εμείς μετρήσαμε ακριβώς ε, το τι γίνεται από την στιγμή της πρώτης υποδοχής. Λέμε εκεί πέρα στις γυναίκες ότι θα πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία. Το άλλο θέμα είναι η πρόσβαση στην υγεία αλλά και σε οτιδήποτε αφορά τον σεβασμό του πολιτισμού της προέλευσης αυτών των ανθρώπων γιατί υπάρχει θέμα και πρόβλημα συνεννόησης παραδείγματο χάρη ας μιλήσουμε για τις ε, γυναίκες οι οποίες υφίστανται σεξουαλικό ακροτηρισμό των γεννητικών οργάνων υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ε, σιωπούν και κάτι άλλο το οποίο επίσης ε, πρέπει να τονίσουμε είναι αυτό το οποίο κάνει η Ιταλία για τις γυναίκες οι οποίες ε, καταγγέλουν ε, ότι έχουν υποστεί βία, λαμβάνουν μια ανθρωπιστική άδεια διαμονής. Κάτι το οποίο νομίζω θα μπορούσαμε να το μοιραστούμε και με άλλα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας η οποία θα πρέπει να συνδεθεί νομίζω και με εκστρατείες ε, ενημέρωσης και σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης αυτών των γυναικών και να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Thank ε, ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που ήμουν τόσο αυστηρός ε, στην τήρηση του χρόνου και δεν είχατε αρκετό χρόνο για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Άννα, ένα λεπτό παρακαλώ, γιατί πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία. Την περασμένη εβδομάδα στην πατρίδα μου την, Πορτο... μου, την Πορτογαλία ένα δίκτυο με ε, δύο, γυναίκες και... δύο άντρες και μία γυναίκα ανακαλύφθηκε ότι κρατούσε 36 γυναίκες διαφορετικές προέλευσης, κυρίως από την Ιγυρία όμως, και αυτό το κύκλωμα χρησιμοποιούσε αυτές τις γυναίκες όχι μόνο για ε, αναγκαστική πορνεία αλλά και για ε, συνουσία χωρίς προστασία και μάλιστα οι γυναίκες αυτές κρατούνταν εχμάλωτες ε, και υφίσταν και ξυλοδαρμό και βιασμό. Και μάλιστα το κύκλωμα αυτό είχε παρακλάτη και σε πολλές άλλες πόλεις. Και μάλιστα κάποια τμήματα ε, ενεργοποιούνται σε Νεγάλη, Γιουνέα, Μπισάο, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Βλέπετε λοιπόν ότι πρόκειται πραγματικά για εγκληματική οργάνωση με τέτοιε εγκληματικέ επιχειρήσει. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βασιλιάδου για το έργο τη και να ρωτήσω σε τι βαθμό εξετάζουμε την εμπορία ανθρώπων από Λιβύη, από Τουρκία και κατά πόσο την εξετάσουμε και υπό αυτό το πρίσμα. Συνάδελφοι, πήγε 12, θα χρησιμοποιήσουμε άλλα 5 λεπτά, ήρθατε για την πληροφορία, αλλά θα καθυστερήσουμε άλλα 5 λεπτά. Ε, και τώρα πια που έχουμε μεγάλο κοινό, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, όπως ήθελε και η κυρία Βασιλιάδου, να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχετε 5 λεπτά, κυρία Βασιλιάδου, για να απαντήσετε. Ξέρουμε ότι θα μπορούσατε να μιλήσετε και περισσότερο. Ε, προσπαθήστε όμω να είστε σύντομοι και να απαντήσετε στα βασικότερα θέματα που τέθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα θα απαντήσω για τα δεδομένα. Για να συνοψίσω και τα σχόλια που ακούστηκαν. Τα δεδομένα εξαρτώνται από, από το τι μας μεταβιβάζουν τα κράτη-μέλη. Εγώ νιώθω λίγο άβολα με τις εκτιμήσεις. Η Eurostat δεν χρησιμοποιεί εκτιμήσεις, ε, ούτε οι άλλες υπηρεσίες μας. Οπότε... Ε, εμπιστεύομαι τα νούμερα που έχουμε. Αυτό που δεν έχουμε είναι ε, ε, επαρκής εντοπισμούς θυμάτων για σεξουαλική εκμετάλλευση, για ε, καταναγκαστική εργασία, για λαθρεμπόριο οργάνων. Θα έπρεπε κανονικά να έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα. Το 2007... Από το, από το 2004 μάλλον οι εκθέσεις μας αναφέρουν ότι ε, δεν αξιοποιούνται όλα τα εργαλεία. Το 2011 είπαμε ότι πρέπει να ε, παρέχεται συνδρομή προς τα θύματα. Επίσης δεν είναι επερκής. Το πρόβλημα δεν είναι η νομοθεσία που μας λείπει, αλλά η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Να πω κάτι για το κυβερνοέγκλημα, κάτι που μας απασχολεί και μας προβληματίζει πάρα πολύ. Επαγρυπνούμε και το παρακολουθούμε πολύ στενά στη συνεργασία με τη Europol. Έχουμε κάνει πολλές επισκέψεις σε χώρες. Ιταλία, Ρουμανία και Ελλάδα επέρχονται και προσπαθούμε να προωθήσουμε τη χρήση κοινών ομάδων διερεύνησης ακόμα και με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων της Ευρωπόλ. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να εξετάσουμε αυτό το θέμα των ε, Ευρωπαίων θυμάτων και χαίρομαι που πολλοί Ευρωβουλευτές επισήμαναν αυτό το ζήτημα. Είναι θεμελιώδους ε, σημασίας αυτό. Και αυτό άλλωστε συμπεριλαμβάνεται και στην έκθεση προόδου μας όπου επίσης επισημαίνουμε βέλτιστες πρακτικές από τα κράτη-μέλη, γνωρίζουμε τη συζήτηση που γίνεται για τις πληροφοριοδότες και την προστασία τους και συμμετέχουμε και εμείς στη διαδικασία αυτή. Και τέλος για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση νομίζω ότι το σημαντικότερο θέμα είναι η δουλειά μου, δουλειά σας να ενημερώσουμε ενημερώσουμε και να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά τα θέματα. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλα, όχι από έλλειψη σοβασμού, αλλά από έλλειψη χρόνου. Θα ήθελα παρόλα αυτά να σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βασιλιάδου, βλέπετε ότι το έργο σας χαίρει μεγάλης εκτίμησης ε, και ε, είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα για κάποια επόμενη έκθεση. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφους που είναι στη συζήτηση. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Είστε όλοι έτοιμοι? Λοιπόν, Ξεκινούμε με την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Έντομα Προστασίας. Ε, Σωράγια Πώς, Τερέζα Χιμένες Μπεστερίλ Μπάριο. Η Σωράγια δεν είναι εδώ. Ε, Τερέζα, θέλεις σύντομα να πάρεις τον, το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω α, απλώς ε, τους και ηγητές για τη συνεργασία μας που ήταν πραγματικά ε, πολύ εύκολη γιατί βρισκόμασταν όλοι στην ίδια γραμμή πλεύσης. Ε, είχαμε μεγάλη σύμπνοια ιδεών. Είμαστε στο πλευρό των θυμάτων, των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και νομίζω ότι ως προς αυτό υπάρχει απόλυτη ομόνια απόψεων και ε, σύμπτωση απόψεων και ευχαριστώ και τη Γραμματεία. Μην ξεχνάτε ότι η οδηγία αυτή ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια με υψηλέ προσδοκίες και τελικά ήταν μια παταγώδη αποτυχία, ε, γιατί δεν ζητήθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα απομάκρυση. Ε, γιατί αυτό που θέλαμε ήταν να προστατεύσουμε τα θύματα και δεν ε, υπήρξαν αιτήματα για τέτοιε εντολέ. Άρα πήγαν όλα στράφη πήγε χαμένη η οδηγία και τώρα προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση και να συμπληρώσουμε το μείζον πρόβλημα που είναι η άγνοια. Θα πρέπει να γνωρίζουν τα θύματα, οι αστυνομικοί, οι δικαστές, την ύπαρξη αυτής της οδηγίας και τη δυνατότητα βελτίωσης της προστασίας που παρέχουμε στα θύματα. Και με την σημερινή ψηφοφορία θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ζητώντας στατιστικά στοιχεία για να δούμε τι συνέβη και Πού οφείλεται μέχρι τώρα αποτυχία. Σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες και για την συμβολή σας. Ευχαριστώ Τερέζα. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 8, πρώτη ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 68. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 69. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 72. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Τροπολογία 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 11, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 85, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τροπολογία 86, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 102. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 102 και 103 σωστά το επισημαίνει στο μας. Δεν έχω κλείσει ακόμη την ψηφοφορία. Τώρα κλείνει και απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 15. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 114. Άρχιτη ψηφοφορία. Ε, τροπολογία, συγγνώμη, έχει συμβαστική. Τέλος ψυχοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 123. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 124 και 125 είναι πανομοιότυπες. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτονται. Τροπολογία 126. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 127. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 128. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 129. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 130 και 133. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 134, 135 ταυτίζονται. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 136, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 137, 138 ταυτίζονται. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 139. Ψηφίστε παρακαλώ αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 144. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 145. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της Εγκρίνεται. 146. Άρχεται ψηφοφορία. Όχι. Καταπίπτει. 147. Υπέρ. Ε, άρχεται ψηφοφορία. 147. Ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 147. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 149. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Απορρίφθηκε η τροπολογία. 151. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 22. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 162-163 ταυτίζονται. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 165 και 100... 165 μόνο. Άρχισε η ψηφοφορία. η ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 167. η ψηφοφορία. η ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 168. η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέ... Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 173. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 174. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 175 ψηφίζουμε. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 176 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. 177, 178 ταυτίζονται. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Α, και οι 179 ταυτίζονται και οι 3. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Τροπολογία 180 και 181 που ταυτίζονται. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Τροπολογία 182. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 183. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχιτη ψηφοφορία. Ε, Πέρα ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 3. Okay, just indicate um, later if you, if just make a record and indicate later. Εντάξει, πείτε το αργότερα λοιπόν. Ε, τροπολογία, συγγνώμη, κλείνουμε, κλείνουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία 3. Στην τροπολογία 3 είμαστε, εντάξει. Λοιπόν, τώρα τελειώνει Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία επί τη τροπολογιστρία. 3. Απορριφθήκε και πάμε στην τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Αγωνία εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ψηφίστε παρακαλώ. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Θεολογικέ αναφορέ. Τροπολογία 7. η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 8. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 12 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 15. Όχι, συγγνώμη, 14. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 18. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 19. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε και εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Συμβαστική 5, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφοφορία ολοκληρώθηκε, εγκρίνεται. Συμβαστική 6, άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 44, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 47 υπέ, ε, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 7 άρχιτη ψηφοφορία. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά τώρα. The vote is closed. εγκρίνεται. 54 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, μια αποχή συγχαρητήρια στις κυρίες Μπεσαρέλ και Πόστ. Τελειώσαμε με την ψηφοφορία συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε στις 2 και μισή για την, με την συνεδρίασή μας για τις διεθνείς επιπτώσεις.